μέχρι την 11η Φεβρουαρίου. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι η γραπτή δήλωση 54 του 2009 για τη μεταφορά των αλόγων για σφαγή της κυρίας Ελίζα Βεθλίν και του κύριου Κάρλ Σλούτερ της, συντονία Συντονίας για τη υπογράφηκε το 24, 24 Φεβρουαρίου του 2010 οπότε με βάση το άρθρο 123 παράγραφος 4 του κανονισμού θα διαβιβαστεί μαζί με τις υπογραφές ε, των συντακτών και των συνυπογραφών των στα πρακτικά της σημερινής συνόδου της και τη συνόδου 25 Φεβρουαρίου του 2010. Ευχαριστούμε τους ε, τρει συντάκτε για την ε, συγγραφή αυτής της γραπτής δήλωσης. Ε, υπέγραψα τη δήλωση. Είναι καλά μαντάτα αυτά που πετύχαμε αρκετές υπογραφές. Ευχαριστώ όλους που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση. Κυρία μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εγώ δεν πρόλαβα να προσυπογράψω αυτή τη γραπτή δήλωση, αλλά είμαι έτοιμος να το πράξω αμέσως. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές με ενημέρωσαν ότι με ισχύ από τη 10η Φεβρουαρίου 2010 η θέση του κυρίου Μισελ Μπαρνιέ θα πληρωθεί από την κυρία Κωνσταντς Λεγκρίπ. Καλωσορίζουμε τη νέα συνάδελφα.